Περνάμε τώρα στην επόμενη έκθεση. Είναι η έκθεση Swinburne σχετικά με την ανάκαμψη και την εξυγίανση για μη πιστοτικά ιδρύματα. Το ρόλο, ε, τον λόγο έχει η συγγήτρια, παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, η οδηγία αυτή αφορά τι συστημικές αδυναμίες που διαπιστώσαμε κατά τη διάρκεια της κρίσης και το θέμα των υποδομών. Προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε τις επιπτώσεις λόγω της έλλειψης ακριβώ νομοθεσία πριν από την κρίση. Το έργο της αποκατάστασης των τραπεζών αφέθηκε στα χέρια των κυβερνήσεων, αλλά δεν έχουμε σταθεροποιήσει τι κρίσιμε υποδομέ τη αγορά. Οι αγορές είναι πολύ περισσότερο αλληλοσυνδεδεμένε και αυτό θα αποδειχθεί, φοβούμε, μια μελλοντική δυναμία των αγορών στο σύνολό του. δούμε τι γίνεται όταν μια τράπεζα καταραίει, αλλά ακόμη περισσότερο τι γίνεται όταν καταραίει ολόκληρη η υποδομή που στηρίζει τι τράπεζε εν γέννη. Αυτό ο κίνδυνο είναι υπαρκτό. Χρειαζόμαστε λοιπόν κεντρικού φορεί διακανονισμών, του CSD, για να αντιμετωπίσουμε ακριβώ τους σχετικού κινδύνους, όχι μόνο των τραπεζών, αλλά και των ασφαλιστικών εταιριών και των εταιριών διαχείριση περιουσιακών στοιχείων. Όλο και περισσότερες συναλλαγέ εκαθαρίζονται κεντρικά. Πολύ περισσότερο από το 2008. Ο όγκος των σχετικών συναλλαγών έχει αυξηθεί εκθετικά και ακόμη περισσότερο θα το πράξει στο μέλλον. Η κεντρική αντισυμβαλόμενοι θα, παίξουν, θα πρέπει να παίξουν ακόμη πιο σημαντικό ρόλο. Επίσης, το ίδιο ισχύει για τον κανονισμό για τις υποδομές των ευρωπαϊκών αγορών, τον κανονισμό ΕΜΙΡ. Έτσι θα εξασφαλίσουμε περισσότερη διαφάνεια στις χρηματοπιστωτικές αγορές. Στην περίπτωση αστοχίας πρέπει οι κεντρικοί ενσημελόμενη να είναι εκεί και να έχουν έτοιμα σχέδια αντιμετώπισης της κατάστασης. Υπό την υποπτία βεβαίω των σχετικών αρχών, οι οποίες θα παρεμβαίνουν όποτε πρέπει. Η εκθέση αυτή τονίζει ότι οι καθημερινές συναλλαγές πρέπει να συνεχίσουν να δημιουργούν κίνητρα για καλή διακυβέρνηση. Έτσι λοιπόν οι κεντρικές τράπεζες θα έχουν το κίνητρο να συμμετέχουν σε κεντρικούς πληστηριασμού και να μην εκαθαρίζουν προϊόντα τα οποία, των οποίων τον κίνδυνο δεν μπορούν να διαχειριστούν. Γιατί στο τέλο έχουμε πελάτε του οποίου ακριβώ πρέπει να προστατεύσουμε γιατί δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν κινδύνου που δεν κατανοούν. Έτσι λοιπόν, εάν κάποιο κεντρικό συνδυασμένο αστοχήσει, πτωχεύσει, έτσι οι τελικοί πελάτε θα είναι προστατευμένοι. Το κεντρικό αυτό όργανο πρέπει όμως να οριστεί και να κοινωθεί. Το Κοινοβούλιο κατέληξε σε ισχυρή συμφωνία προ την κατεύθυνση αυτή. Ότι πρέπει δηλαδή να υπάρχουν μέτρα μεταξύ των ε, κεντρικών αντισυμβαλωμένων. Υπό την υποπτία πάντοτε της κεντρικής αρμόδιας αρχής. Στην περίπτωση που κινδυνεύσουν τα περιουσιακά στοιχεία του τελικού πελάτη, υπάρχει λύση υπό την οπτία λοιπόν της κεντρικής αρχής. Πρέπει εμείς να φροντίσουμε ότι υπάρχουν από σήμερα συστήματα και ότι οι κεντρικοί ενσυμβαλόμενοι θα, θα εξαντλήσουν πρώτα τις δικές τους δυνατότητες πριν να παρεύουν στα περιοχικά στοιχεία του άλλου μέρου. Εάν ο κεντρικό συνδυσφαλόμενο υποχρεούται από την αρχή να χρησιμοποιήσει τα δικά του περιουσιακά στοιχεία, τότε βεβαίω θα έχει κανένα κίνδυνο να λειτουργήσει. Γι' αυτό λέω ότι δεν πρέπει να θίγονται τα συγκεκριμένα περιουσιακά στοιχεία. Όλα αυτά προκύπτουν από την προσπάθειά μα να βάλουμε τάξη στην αγορά. Ο τριμερή διάλογο προχωρεί. Στόχος όλων μας είναι, επαναλαμβάνω, να παράσχουμε λύσεις στην περίπτωση μιας γενικότερης κατάρρευσης. Ευχαριστώ. Δεν βλέπω κανένα να, λάβει το, να θέλει να λάβει το λόγο στην οφθαλμοσυλληπτική διαδικασία. Θα δώσω αμέσως το λόγο στην Επίτροπο κυρία Ρέντιν. Κυρία Πρόεδρε, θέλω να ευχαριστήσω την κύρια Σουάινμπερν για μια θαυμάσια έκθεση. Είναι γεγονός ότι το ρυθμιστικό πλαίσιο στον τομέα αυτό ευθυγραμμίζεται με τις διεθνείς δεσμεύσεις που ελήφθησαν σε επίπεδο των G20 για να βελτιωθεί η λειτουργία των χρηματοπιστωτικών αγορών και να αποτρέψει το να πρέπει οι φορολογούμενοι να φέρουν το κόστος της ε, αστοχίας των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Χαιρετίζουμε τη συμβολή αυτής της έκθεσης σε αυτό το σημαντικό ζήτημα επί τη βάση των δικών μας διαβουλεύσεων, επί τη βάση των διεθνών ε, εργασιών που έχει γίνει από το Διεθνές ε, Συμβούλιο συστημικής ασφάλειας θέλουμε να δημιουργήσουμε τους κατάλληλους, τα κατάλληλα εργαλεία για την ε, ανάκαμψη και την επίλυση συστημικών φορέων. Λόγω του συστημικού φορέα αυτοί οι φορείς θα αποκτήσουν ακόμα μεγαλύτερη σημασία εφόσον το Συστημικό Συμβούλιο θέλει να εφαρμόσει τη μεταφορά από την, ε, από την εκτός αγορά στην σε αγορά επί τη βάση κεντρικών αντισυμβαλωμένων. Θα πρέπει λοιπόν να κάνουμε τις απαραίτητες προσπάθειες για να εφαρμοστούν οι πιο στεναροί εποπτικοί κανόνες ώστε να υπάρξει και η κατάλληλη ρύθμιση των κεντρικών αντισυμβαλωμένων και να υπάρξουν οι προτάσεις για την ανάκαμψη και την επίλυσή τους επί τη βάση των διεθνών εργασιών που έχουν γίνει. Εμείς τονίζουμε τη σημασία, χαιρετίζουμε τη σημασία μάλλον που έχει δοθεί σε μερικά από τα κύρια θέματα που αφορούν την ανάκαμψη και την επίλυση των κεντρικών αντισυμβαλωμένων, πραγματικά χάρη μηχανισμοί για να αντιμετωπιστούν οι εποπτικές απώλειες και οι συμβατικές ρυθμίσεις για κάτι τέτοιο θα πρέπει να είναι διαφανείς και αποτελεσματικές διότι μας ενδιαφέρει να ατηρηθεί η συνέχεια του ρόλου των κεντρικών αντισυμβαλωμένων. Βέβαια αυτή η συνέχεια δεν πρέπει να γίνει με έναν τρόπο ο οποίος πλήττει τους χρήστες των ε, κεντρικών αντισυμβαλωμένων ή οδηγεί σε ηθικό κίνδυνο. Η Κομισιόν λαμβάνει υπόψη όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία αναφέρονται στην έκθεση και θα τα λάβει υπόψη όταν δώσει τη δική της πρόταση για τα θέματα αυτά. Ευχαριστώ πολύ. Ολοκληρώθηκε η συζήτηση. Η ψηφοφορία θα λάβει χώρα αύριο στις 11.30. Siamo in attesa dell'onorevole Nibler e quindi dobbiamo attendere qualche secondo. Αναμένουμε τώρα την κυρία Νίμπλερ, η οποία είναι καθοδόν.